και έχω λάβει από το Συμβούλιο θέσει σε πρώτη ανάγνωση καθώς και τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτησή τους και τις αντίστοιχες θέσεις της Επιτροπής. Θα καταχωρηθούν οι τίτλοι στα πρακτικά ε, και ε, ξεκινάει η προθεσμία τριών μηνών για το Κοινοβούλιο από αύριο 28 Φεβρουαρίου του 2014. Και τώρα περνώ στις επεξηγήσεις ψήφου για τις προφορίες που δεξήφθησαν και έχω πρώτα την έκθεση λένε